Dear colleagues, dear Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ας έλθουμε στην απογευματινή συνεδρίαση και πριν να αρχίσουμε την ακρόαση για την διαθεσμική συμφωνία για μια καλύτερη νομοθεσία, ας μου επιτρέψετε να σας ανακοινώσω τις αποφάσεις των συντονιστών της Νομικής Επιτροπής σχετικά με τους διορισμούς εισηγητών. Φεράρα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Φλόριαν Φίλιππον σε σχέση με δικαστική έρευνα. Η κυρία Χάουταλα θα οριστεί η συγγήτρια για, σχετικά με νέο Έτοιμα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Τσέσλαβ Σικέρσκη σε συνδυασμό με παλαιότερη υπόθεση ώστε θα χρειαστεί μονάχα μια ακρόαση. Η κ. Χάουταλα επίσης θα οριστεί η συγγήτρια γνωμοδοτήσεως για την εφαρμογή της ε, συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών ή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών μάλλον για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και, με την, ε, και σε σχέση με την ε, Επιτροπή UNCPR. Χρειάζεται ειδική έγκριση για να συνταχθεί η γνωμοδότηση αυτή για την οικονομική διαχείριση και την ασφάλεια για υπεράκτιες επιχειρήσεις εξόριξης αερίου σε σχέση και με την απόφαση 2013 οι συντονιστές μάλλον συμφώνησαν να διεξαχθεί εργαστήρι μαζί με εθνικά κοινοβούλια το Γενάρη του 2016 για τις δύο προτάσεις αφενός για την επιγραμμική πώληση ε, αγαθών και για την, την επιγραμμική ε, διακίνηση ε, περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επίσης οι συντονιστές αποφάσισαν οι προφορικές ερωτήσεις για την προστασία των παιδιών διαμεθοριακά στην Ευρώπη θα αρχίσουν οι εργασίες δηλαδή από την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου 2015. Επίσης οι συντονιστές συμφώνησαν να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής για τον Νοέμβριο 12 Νοεμβρίου 2015 δηλαδή, το ζήτημα γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων με στόχο να ακούσουμε έναν εμπειρογνώμονα από τον ΟΟΣΑ και να προσκληθεί η Βολουξεμβουργική Προεδρία και η Μελλοντική Ολλανδική Προεδρία και θα προσκληθούν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών. Επίσης συμφώνησαν οι συντονιστές να θέσουν προφορική ερώτηση για το ίδιο θέμα που ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί, άρα θα γίνει γραπτός αυτό η διατύπωσή της. Και οι συντονιστές συμφώνησαν να διοργανώσουν εκδήλωση στο επόμενο έτος όπου η Συμβουλευτική Επιτροπή για την μεταρρύθμιση του πολιτικού τομέα, του μη στρατιωτικού τομέα στην, Ουκρανία, στην Ουκρανία με συμμετοχή και της Ουκρανικής και της Ευρωπαϊκής πλευράς όπου θα προσκληθούν οι εκπρόσωποι τους. Και τέλος η κυρία Ντελβό θα οριστεί πλήρες μέλος, η κυρία Κομοντίνη Κάτσα και ο κύριος Άντερσον αναπληρωματικά μέλη της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Απασχολήσεως για τις επιπτώσεις στην ε, ενιαία αγορά της ψηφιοποίησης, των, της ρομποτικής και της τεχνητής ευφυΐας. Αυτά ε, συναποτελούν τις αποφάσεις των συντονιστών μας και τώρα θα ήθελα να απευθύνω το καλώς ορίσατε ε, σε όλες και όλους εσάς για το πρώτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης που διεξάγεται μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών και η κυρία Βίπνερ που είναι η πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, της Πραγματικής Επιτροπής βεβαίως, θα ήθελα τώρα να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την Συνταγματική Επιτροπή δεν έχουμε ομιλητές, άρα με την ευκαιρία αυτή θα θέσω και ορισμένα ουσιώδη θέματα. Θα γνωρίζετε ότι η τρέχουσα ε, διαθεσμική συμφωνία για βελτίωση νομοθεσίας χρονολογείται το 2003. Ωραίο είναι αυτό βέβαια, ωραία ημερομηνία, ωραία χρονολογία μάλλον αυτή, αλλά τότε η Ευρώπη ήταν πολύ διαφορετική. Ήταν δηλαδή και πριν από τη μεγάλη διεύρυνση που έγινε αργότερα μετά από αυτό, αλλά και πριν από την κρίση η οποία έχει ξεκινήσει πολλές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ε, όπου εμπλουτίστηκε και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων. Επομένως, τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλές και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και γι' αυτό είναι σωστό που οι δύο επιτροπές μας εγκύπτουν στην Διαθεσμική Συμφωνία για την Βελτίωση Νομοθεσίας και αυτή η Διαθεσμική Συμφωνία να επανεξεταστεί σε βάθος, πράγμα το οποίο έχει ζητήσει άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα κατ' επανάληψη έχει ζητήσει αναθεώρηση της ε, εν λόγω συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή εγκύπτει σε θέματα που έχουν θεμελιώδη σημασία για μας και τα περισσότερα μάλιστα για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ο συνάδελφος Σφόμποντα και εγώ δεχθήκαμε το γεγονό ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μέσα στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι οι δυο επιτροπές νομικών και συνταγματικών θεμάτων δηλαδή παίζουν σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να ε, ενταχθούν και αυτές μέσα στην διαδικασία όσο γίνεται περισσότερο. Μάλιστα έχουμε συντάξει έγγραφα που παρουσιάζουν τις απόψεις των επιτροπών μας. Ο Πάουλ Σόβοντα και η νομική επιτροπή βεβαίως είναι η κατεξοχήν μάλλον αρμόδια επιτροπή, αλλά βεβαίως και η δική μας επιτροπή των συνταγματικών δηλαδή διαθέτει και αυτή αρμοδιότητες για διαθεσμικά θέματα, για την εφαρμογή των συνθήκων και για την αξιολόγηση της λειτουργίας των συνθήκων. Επίσης είμαστε αρμόδιοι και για ορισμένες λεπτομερείς πτυχές που γίνονται αντικείμενο χειρισμού μέσα σε αυτά τα πλαίσια της διαθεσμικής συμφωνίας όπως βελτιωμένη συνεργασία στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας και ιδίως ό,τι αφορά το διαθεσμικό προγραμματισμό και ιδίω πολιετή προγραμματισμό που είναι σημαντικός για μας και από τις ακροάσεις που έχουμε ήδη διεξαγάγει μαζί με τον Γκίφερ Χόφστατ που είναι ο ε, κύριος διαπραγματευτής για τη συμφωνία αυτή βλέπουμε ότι η συζήτηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων περιστρέφεται γύρω από μια συμφωνία ενίσχυσης του διαθεσμικού προγραμματισμού και μιας καλύτερης διασύνδεσης του πολιετούς προγραμματισμού και σχεδιασμού. Στην ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ είμαστε υπεύθυνε και για την παρακολούθηση της διαθεσμικής ισορροπίας μέσα στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων των αρμοδιοτήτων δηλαδή των διαφόρων θεσμικών οργάνων και ιδίω όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών. Θα θυμάστε ότι επί δεκαετίες ολόκληρες θα έλεγα υπήρχε ένα είδος υποφόσκουσας σύγκρουσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με το σε ποιον ε, υπόκειται στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν. Και έχουμε και ένα ρόλο να παίξουμε και για άλλες θεσμικές πάγιες αρχές όπως διαφάνεια, όπως ε, η φιλικότητα προς τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και μιας σημαντικής διάστασης βέβαια της νέας συμφωνίας και καμιά φορά οι αρμοδιότητες μας επικαλύπτονται με αυτές τις νομικές επιτροπές, όπως η φροντίδα για την νομιμότητα, για την βελτίωση της νομοθεσίας, για το κράτος δικαίου. Άρα οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και για θέματα επικουρικότητας, αναλογικότητας, τα οποία είναι πολύ επίκαιρα, θα θέλαμε επίσης να δούμε αυτήν την βελτίωση της νομοθεσίας να θεωρηθεί όχι απλά ως λιγότερη νομοθεσία, διότι αυτός ο στόχος της λιγότερης νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει και σε δυσκολίες. Δεν είναι, το μόνο αντικείμενο δεν μπορεί να είναι να αποσύρονται νομοθετικές προτάσεις, πρέπει να προτείνονται και εναλλακτικέ δυνατότητες, εναλλακτικέ νομοθετικές δυνατότητες. Να μειώνεται βεβαίω και το γραφειοκρατικό βάρος. Και όταν υποβάλλουμε προτάσεις, αυτό πρέπει να γίνεται μέσα σε δημοκρατική διαδικασία. Η νομοθεσία αυτή είναι αναγκαία για σημαντικά θέματα, για την βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, για την βελτίωση της λειτουργίας της διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για την καλύτερη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και για την σφυριλάτηση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε και οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές και το Κοινοβούλιο να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά και η ουσία των προσπάθειών αυτών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη νέα δυνατότητα κοινή δράσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων βελτίωση της νομοθεσίας, βελτίωση της ποιότητας, λιγότερο διεισδυτική, βελτίωση της διαφάνειας, καλύτερα ισορροπημένη από μια αρχή από τους νομοθέτες. Όλα αυτά διότι θεωρούμε ότι η βελτιωμένη νομοθετική διαδικασία θα βρει απήχηση στους πολίτες και θα προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω και τις απόψεις που με διακατέχουν σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες μας από την διαδικασία αυτή. Θα θέλαμε να δείξουμε ότι τα κοινοβούλια αν συνεργάζονται θέλουμε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή γιατί αυτό θα οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χίπνερ. Λέει ο πρόεδρος Φόβοντα, πριν δώσω το λόγο στον αξιότιμο κύριο Καρύμ να Πότε εξή, Στην αίθουσα παρευρίσκεται αντιπροσωπεία ε, αξιωματούχων της Ιταλικής Γερουσίας. Σας απευθύνω ε, θερμό, εγκάρδιο, καλώς ορίσατε. Benvenuti, είναι η μόνη λέξη που μου έρχεται τώρα αυτά Ιταλικά. Και δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε προσκαλέσει και προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την παρουσία του κύριου Τίμπερμαντς όπως και του κυρίου Φερχόστατ στην ακρόαση. Δυστυχώς τα πρόσωπα αυτά δεν μπόρεσαν να είναι παρόντα σήμερα, άρα θα κάνουμε την ακρόαση χωρίς αυτούς. Ε, ο κύριος Καρίν θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά σας είμαι υπόχρεος που μου δίνετε αυτή τη στιγμή το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα εισαγωγικά είπατε κι εσείς και η κυρία Κούνα ως πρόεδρος ε, της Σχετικής Επιτροπής. Ευχαριστώ που, ε, για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Θίξατε το θέμα που ήθελα να θέσω κι εγώ, γιατί σκεφτήκαμε να οργανώσουμε αυτή αυτή την ε, ακρόαση σκεπτόμενοι ότι θα ακούσουμε απόψεις από τον, σχετικό, τον αρμόδιο επίτροπο και από τον κύριο, από τον κύριο Τίντερ μας και από τον κύριο Περχόφστατα. Ακούσαμε ότι η θέση του είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις ε, ε, διαθεσμικές συμφωνίες και πραγματικά δίχω τον κύριο Βερχόφσταρ και τον κύριο Τίντερ μας τα έλεγα ότι δεν είναι συζήτηση στην ουσία. Μεταξύ μα τα μιλάμε, μόνοι μα τα λέμε, μόνοι μα θα τα ακούμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφάνειας, διαφάνειας διαδικασιών, πολύ φοβάμαι και δεν είμαι ο μόνος που το φοβάται ότι Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που απαιτούν μία απάντηση πριν να περάσουμε σε μία φάση όπου θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επιθεμάτων ουσίας. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ακρόαση, το γεγονός ότι ο κύριος Τίντερμας και ο κύριος Βερχόφστατ υψηλή ε, αξιωματούχοι, τον ένα έχουμε καταλάβει τι κάνει, για τον άλλο τα πράγματα είναι κάπως ασαφή. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου δυνητικά θα τους, θα τους δώσουμε ασαφή στοιχεία γιατί στην ουσία ε, σε ό,τι αφορά την, ε, τη δημοκρατική κάλυψη είναι γυμνή. Το παρελθόν ήταν μια διαδικασία που δεν μας κάλύπτε ε, πουδενή. Τώρα είναι μια διαδικασία την οποία θεωρούμε απλώς απαράδεκτη. Εμείς ήρθαμε εδώ θεωρώντας ότι δύο αυτοί κύριοι θα έρθουν εδώ ενώπιον μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Τώρα πραγματικά δεν έχω καμία άλλη επιλογή παρά το να αφήσουμε κατά μέρος αυτή την ακρόαση και να γίνει όταν τα, οι δύο ε, αυτοί οι αξιωματούχοι έρθουν καταδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα έλεγα ότι η Επιτροπή αυτή δεν θα τους δώσει φίλος για να καλύψουν τη γύμνια τους όσο δεν εμφανίζονται μπροστά μας. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η ε, κυρία Νίπλερ. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Καρίμ. Δεν μπορώ να αποδειχθώ την διαδικασία αυτή. Υπενθυμίζω ότι επί μήνε έχουμε ασχοληθεί με την βελτίωση της νομοθεσίας εκεί. Η κυρία Κάουφμαν είχε συντάξει έκθεση, είχαμε καταθέσει τροπολογίε. τη συζητήσαμε, τον, ψηφίσαμε την έκθεση αυτή και μετά όπω και πολλέ και πολλοί συνάδελφοι διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι η έκθεση δεν καταλήγει στην Ολομέλεια για ψήφιση, διότι, αυτό ακούμε, λόγω της ε, συζήτησης για την διαθεσμική συμφωνία αναστέλλεται η πορεία της έκθεσης. Εμένα μου φαίνεται ασυνήθις αυτή η διαδικασία και μαθαίνω ότι η συζήτηση με τους κύριους Φερχόφστατ και Τίμερμανς υποτίθεται θα γινόταν, θα είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τα ίδια πράγματα τώρα ενώπιόν τους, αλλά βεβαίως σήμερα λείπουν οι δύο αυτοί βασικοί συνομιλητές. Ε, όπως είπα και πριν, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καρίμ και εκφράζω με έμφαση την παράκληση. Ο κύριος Ερχόστατ, στο κάτω της γραφής, διαπραγματεύεται για λογαριασμό του Κοινοβουλίου. Ας εμφανιστεί ενώπιον του ε, κοινοβουλίου εμφανιστεί ενώπιον της Νομικής Επιτροπής. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με τον συναδελφό μου. Ίσως λοιπόν έχει νόημα όντως η συζήτηση που προτιθέμεθα να κάνουμε σήμερα να αναβληθεί για ε, κάποια άλλη ημερομηνία όπου να είναι δυνατόν τα πρόσωπα αυτά να είναι παρόντα. Mrs. yes. Κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ. Συμφωνώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συμφωνήσω. Μιλούμε για βελτίωση της νομοθεσίας, βελτιωμένη νομοθεσία. Έχουμε μπροστά μας ένα παράδειγμα που στην ουσία είναι χειρότερη νομοθεσία. Η παρούσα επιτροπή που είναι αρμοδία και βεβαίως και η Επιτροπή Συνταγματικών δεν έχω παρά να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου. Έχουμε συντάξει έκθεση, έχουμε εκπονήσει έκθεση η οποία είναι έτοιμη. Το μόνο που μπορώ να συμπληρώσω είναι ότι έχουμε την έκθεση εφόσον εκπονείται άλλη έκθεση με διαφορετικό τίτλο στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, περιέχει όμως παρόμοια θέματα με αυτά της, κυρίας, της εκθέσεως της κυρίας Κάουφμαν και αυτή η δεύτερη έκθεση πάει να φτάσει στην Ολομέλεια. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας κάτι πάει στραβά. Ότι χρειάζεται σύναψη διαθεσμικής συμφωνίας αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως πολλά τα οποία εμπίπτουν στην, στις αρμοδιότητες των αρμοδίων επιτροπών δεν προωθούνται επαρκώς. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου και όχι απλά να παρακαλέσω τους δύο αυτούς συνομιλητές που αναφέρατε, αλλά να τους ζητήσω να έλθουν, να απαιτήσω να έρθουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα. Και πιστεύω ότι η άρνηση των δύο ανδρών είναι δείγμα αλαζονίας, είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε μία αρχή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα βροντερό μήνυμα και στους δύο, να τους πούμε ότι δεν δεχόμαστε αυτή την άρνηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Τους καλέσαμε, θεωρήσαμε ότι θα υπάρχει μια καλή ανταλλαγή απόψεων μαζί τους σχετικά με το τι σημαίνει καλό ε, ε, εύρυθμοι κανονισμοί. Ε, θα ήθελα... Η κυρία Φαν Μπούσετ, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω αυτό το θέμα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ο κύριος Φερχόφστατε ενδιαφέρεται πάντοτε για τη διαφάνεια και διαπραγματεύεται εξ του Κοινοβουλίου τη, διαθεσμική τη διοργανική συμφωνία. Ίσως μόνο το 1% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζει τι ακριβώς διαπραγματεύεται και δεν έχει κανένα εντολή γιατί δεν μας μίλησε ποτέ και δεν ξέρουμε τι διαπραγματεύεται εξ ονόματός μας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ε, ντροπή οι τρόποι που έχουν πάρει τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κατά βάση συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ωστόσο. Δεν είμαστε μόνο μεταξύ μας. Έχουμε και έναν ε, επίτιμο προσκεκλημένο εδώ, τον κύριο Ρόμπινσον, ε, ερευνητή στο Ινστιτούτο Προηγμένων Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε την ε, αναβολή της ακρόασης ή να ακούσουμε τουλάχιστον τον προσκεκλημένο μας από το Λονδίνο, να κάνει την παρουσίασή του και μετά να ψηφίσουμε την ε, ε, αναβολή της ακρόασης. Ε, τι πιστεύετε κύριε Καρίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων στην Χάιντι Χάουτλα που έθεσε το ζήτημα αυτό και έχω πρόταση και θα ήθελα να τεθεί προς ψήφιση πριν προχωρήσουμε, το εξής δηλαδή. Ο προσκεκλημένος μας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να μιλήσει από τις 3 και 10 μέχρι τις 3 και 25, ο κύριος William Robinson, να κάνει την παρουσίασή του και αμέσως μετά, χωρίς να έχουμε ερωτήσεις προς τον κύριο Ρόμπινσον και χωρίς να γίνει υπεραιτέρω ε, διάλογος, να ε, διακοπεί η ακρόαση, να ανασταλεί. Και το προτείνω αυτό για να εκφράσω το σεβασμό μου στο γεγονός ότι ο κύριος Ρόμπινσον έχει ε, κάνει τεράστια προσπάθεια, έχει κάνει τεράστια δουλειά για να είναι μαζί μας σήμερα και να παραστεί στη διαδικασία. Και θα είχε τύχει τρομακτικού σεβασμού ε, αν δεν είχαμε αυτούς τους δύο τους οποίους όλοι γνωρίζετε εδώ. Ε, λοιπόν Πρόεδρε αυτό να ψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ο κύριος Φερχόφστατ είχε κάποια προβλήματα με την ατζέντα του σήμερα, με το πρόγραμμά του δηλαδή. Είναι στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ενδεχομένως. Δεν είναι ότι αρνήθηκε να παραστεί δήλωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα. Και εγώ είμαι υπέρ του να ψηφίσουμε την αναβολή της ακρόασης σε μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να ε, εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής οι δύο αυτοί κύριοι. Αυτή δεν είναι η πρόταση αν τα κατάλαβα καλά. Επομένως προτείνεται, κύριε Καρίμη να, ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ρόμπισον και μετά να ψηφίσουμε. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Καρίμη. Να ψηφίσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Ρόμπισον και να λήξει η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόταση. Ποιος είναι υπέρ αυτού? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαφέστατα τούτων λεχθέντων και τούτων ε, γενόντων. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλιαμ Ρόμπινσον, τον οποίο σας έχω ήδη παρουσιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο για αυτό το ζήτημα και συμφωνώ με την κυρία Χιούμπνερ. Είναι ένα ζήτημα θεμελιωδός σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει κανείς να το πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά. Εδώ και αρκετό καιρό επιχειρηματολογώ λέγοντας ότι τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην ομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επανεξετάσουν την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει σε αυτή την ομοπαρασκευαστική διαδικασία. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω τη νέα διαθεσμική διοργανική συμφωνία και νόμιζα και ήλπιζα ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως στην πραγματικότητα το κείμενο που προπαρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι και τόσο διαφορετικό από αυτό που είχε παρουσιάσει το 2003 τη Συμφωνία για την Καλύτερη Παρασκευή Νομοθεσίας σε εποχές πολύ διαφορετικές. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια χαμένη ευκαιρία. Χρειάζεται μια πιο τολμηρή προσέγγιση. Και θα έλεγα και θα πρότεινα η νέα αυτή πιο τολμηρή προσέγγιση να έχει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, η νομοθετική αρχή να έχει την ιδιοκτησία ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ownership. Δεύτερον, ε, τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται σε αυτή την νομοπαρασκευαστική διαδικασία να θεσπίσουν ένα πλαίσιο ε, κανονιστικού έργου το οποίο να ταιριάζει στο σκοπό αυτό, να είναι περιεκτικό, συνολικό αλλά και προσβάσιμο. Και τρίτον, για να διασφαλίσουμε συστηματικά ότι αυτό το σχήμα δουλεύει, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδους, μια από κοινού εποπτεία και θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες στο κάθε ένα από αυτά τα τρία στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημοκρατικό σύστημα και διέπεται από το κράτος δικαίου βάσει των συνθήκων οι οποίες επιβάλλουν το άνοιγμα, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ένα τέτοιο σύστημα, κατά την άποψή μου, είναι προφανές ότι η νομοθετική αρχή αυτή αυτή, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι τα θεσμικά όργανα που θα πρέπει να θεσπίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, σε συμφωνία βεβαίω με, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζοντας το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπει κανεί σκιέ και αποχρώσεις της παλιάς τεχνοκρατικής προσέγγισης που είχαμε υιοθετήσει στα πολύ παλιά χρόνια, όπου όλα ήταν εξαιρετικά τεχνικά και τεχνοκρατικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την σιδερένια λαβή, το ισχυρό χέρι που κρατούσε ε, ε, τα πράγματα, αν θέλετε. Για παράδειγμα, στην αξιολόγηση αντικτύπου, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφήστε το σε εμά. Έχουμε τη δική μα προσέγγιση για το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διαμορφώσουν τη δική του προσέγγιση με βάση τη δική μα. Διαφωνώ. Για την απλούστευση, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί έχουμε το δικό μα πρόγραμμα απλούστευση και θα πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να το υιοθετήσουν ω βάση εργασία. Δεν συμφωνώ. Η νομοθετική αρχή είναι αυτή που θα πρέπει να πει τι είδους πρόγραμμα απλούστευσης επιθυμεί και βούλεται. Επομένως, η νομοθετική αρχή θα πρέπει να πάρει τα ημνία σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μαζί θα πρέπει να καθορίσουν τις βάσεις. Οι βάσεις αυτές θα πρέπει να ε, καλύπτουν τις τεχνικές πτυχές των θεμάτων. Πάντοτε θα υπάρξει πολιτική διαδικασία η οποία πάντοτε θα είναι και περίπλοκη. Ωστόσο, πολλά, πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα είναι ζητήματα που χρήζουν κοινή συμφωνία και βασικών κανόνων τεχνιδιών. Για παράδειγμα, σχεδιασμό, προγραμματισμό, διαβούλευση, αξιολόγηση αντικτύπου, κανόνε για τη διατύπωση, κανόνε για τη δημοσίευση και διάδοση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενημέρωση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα και μπορούν να υπόκεινται σε βασικού κανόνε και να ισχύουν βέβαια οι, ίδιοι βασικοί κανόνες και στις πράξεις, στις νομοθετικές ή άλλες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι ένα μοσαϊκό συγκεχημένο παλιό σαν μια ε, ε, ε, κουρελού πλεγμένη από πολλά και διαφορετικά κομμάτια υφάσματος τα οποία είναι μάλιστα και φθαρμένα. Άλλοι κανόνες βρίσκονται στις συνθήκες, άλλοι βρίσκονται στους κανονισμούς. Π.χ. έχουμε ένα κανόνα για τα χρονικά όρια που βρίσκεται σε έναν κανονισμό του 1971. Υπάρχουν και οι κανόνες, οι διαδικαστικοί και οι εσωτερικοί κανονισμοί για το πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν διαθεσμικές ή διοργανικές συμφωνίες, τέσσερις. Υπάρχουν κοινέ δηλώσεις, τρεις. Και υπάρχει και μια συμφωνία πλαίσιο. Ε, αναρρύθμιτες κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια. Κάποια είναι δημόσια και δημοσιευμένα, κάποια άλλα όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Εγώ θα προτιμα ότι θα ήταν καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές αν ήταν κοινέ. Μετά έχουμε ε, ε, ε, διάφορα κείμενα για καλύτερη νομοθεσία, για έξυπνη νομοθεσία, για πιο ισχνή και λεπτή και ευέλικτη νομοθεσία. Μετά η καλύτερη έγινε πιο έξυπνη και αυτό υποτίθεται ότι είναι ακόμα καλύτερο και από το καλό. Και τώρα η πρόταση μας κάνει να επιστρέφουμε στο better regulation, πιο καλύτερη νομοθεσία πολύ απλά, τελεία και παύλα. Ποιος, ξέρει τι συνεπάγονται όλα αυτά. Και υπάρχει και πληθώρα ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε τη διαδικτυακή ε, ε, τοποθεσία, τη διστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταλάβετε πόσες πολλές είναι αυτές οι ανακοινώσεις. Και το πρόβλημα ε, με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε εάν απλά συνυπάρχουν ή αν υπερτερούν οι πλέον πρόσφατες σε σχέση με τις παλαιότερες. Συνεχώς έρχονται και νέοι κανόνες. Και μετά υπάρχουν τα SWD, τα περιβόητα, τα έγγραφα εργασίας του προσωπικού, τα οποία όμως πρέπει να μεταφραστούν και αν δεν έχουν μεταφραστεί δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλοί κανόνες είναι ε, απαξιωμένοι, είναι παλιοί. Το είπε και η κυρία Χιούμπνερ. Η Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία υιοθετήθηκε το 2003, οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τελείως διαφορετική. Οι κανόνες για την κωδικοποίηση είναι του 1994. Οι κανόνες για το recasting, για την αναδιατύπωση και την συγχώνευση της νομοθεσίας είναι του 2002. Και οι κανόνες για τη σύνταξη της νομοθεσίας υιοθετηθήκαν το 98 με την ε, διαθεσμική διοργανική συμφωνία. Είναι δυνατόν κανόνες του 98 να αντικατοπτρίζουν σημερινές ανάγκες. Εγώ θεωρώ πως όχι. Και αρκεί να εξετάσει κανείς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία και βλέπει ότι υπάρχουν εκεί πολλές υποδείξεις και προτάσεις για τις αρχές που πρέπει να διέπουν την σύνταξη, την διατύπωση της νομοθεσίας και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Πολλά παραδείγματα στην πρόταση της Επιτροπής έχουν να κάνουν με τη διατύπωση, το προαπαιτούμενο αξιολόγησης, εποπτείας, αποφυγής της ανάλογου κόστους, αποφυγής κανόνων που είναι δύσκολοι ή αδύνατοι στην εφαρμογή τους. Όλα αυτά υπάρχουν και σε κείμενα του 98. Θα πρότεινα λοιπόν ε, την εξή παραδοχή. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι παλιό, είναι απαξιωμένο, αλλά είναι και ατελές. Ε, ταιριάζουν όλοι αυτοί οι κανόνε στο σκοπό ε, που υποτίθεται ότι επιδιώκουν να επιτύχουν. Και θα έλεγα ότι Μία νέα προσέγγιση είναι αυτό που μας χρειάζεται, να έχουμε όλους τους κανόνες σε ένα και μόνο μέρος. Η νομοθετική αρχή, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίσει, να θεσπίσει όλους τους βασικούς κανόνες σε μια διαθεσμική συμφωνία για την ε, νομοθετική διαδικασία και οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τα βασικά και μετά να έχουμε ε, δευτερογενή κείμενα με περισσότερες λεπτομέρειες και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα υλοποιηθούν τα σχετικά δευτερογενή κείμενα με τις λεπτομέρειες. Πάντοτε ε, με την οπτική γωνία της διαφάνειας. Το θέμα είναι ο καθένας να καταλαβαίνει πολύ καλά το ρόλο του και τους κανόνες ε, τους οποίους πρέπει να υπακούσει. Το ευρωπαϊκό σύστημα βασίζεται πάρα πολύ στους κανόνες γιατί εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων εμπλέκονται στην ομοπαρασκευαστική διαδικασία στα τρία θεσμικά όργανα. Άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια θα έλεγα, από διαφορετικές ιστορικές ή πολιτιστικές διαδρομές και δεν είναι μόνο ειδικοί στην νομοθεσία αλλά έχουν και άλλε εξειδικεύσεις στα προσόντα τους. Επομένως δεν έχουν και ειδική ε, εκπαίδευση στα νομοθετικά ε, θέματα και το γνωρίζω γιατί εγώ είμαι εκπαιδευτής σε σχέση με αυτά. Αλλά ακόμα και αν είναι ε, εκπαιδευμένοι ξέρουν μόνο το πεδίο και το τομέα στο οποίο είναι ειδικοί. Π.χ. Ε, αν κάποιο είναι ειδικό στην αξιολόγηση αντικτύπου, δεν ξέρει καθόλου για κανόνε διατύπωση και σύνταξη νομοθεσία και το αντίστροφο ισχύει. Και μετά πρέπει όλα να μεταφραστούν και οι μεταφραστέ δυσκολεύονται ιδιαίτερω να βρουν μια επισκόπηση όλων των κανόνων που ισχύουν. Επομένω, θεωρώ ότι θα βοηθηθούν και οι αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, τα θεσμικά όργανα αυτά καθεαυτά και θα ενισχυθεί η διαφάνεια, αλλά σύν τη άλλη και οι πολίτε και οι επιχειρήσει θα μπορούν μπορούν όλο και πιο εύκολα να έχουν μια ε, επισκόπηση και μια σύνοψη όλων των κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο αυτή τη χρονιά η Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων δήλωσε και παραθέτω τα εξή. Ο μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων δεν παρέχει επαρκή ευκρίνεια, σαφήνεια, διαφάνεια ω προ του σκοπού ε, των μέτρων και θα πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα κείμενα καλύτερα. Και εγώ αυτό πιστεύω και το λέω. Και ο Ομπουτσμαν, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, έχει πει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε, επιχειρήσει, οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν κάθε στάδιο της νομοπαρασκευαστική διαδικασίας και να κατανοούν πώς οι διαπραγματευτέ φτάνουν στο τελικό σημείο. Το Κοινοβουλίο, η Επιτροπή, όλοι έχουν ενδιαφέρον το Συμβούλιο να νομοθετηθούν όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά να νομοθετούν για να κερδίσουν την ε, δημόσια εμπιστοσύνη. Επομένω εγώ ε, προτείνω ένα σαφέ πλαίσιο των κανόνων του οι οποίοι θα διέπουν τα τρία θεσμικά όργανα και αυτό είναι το πιο ταιριαστό για να μην ε, απολέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την εμπιστοσύνη του κοινού. Δεν αρκεί όμως να εγκρίνουμε απλά ένα σετ, ένα, μια σειρά βασικών κανόνων, όσο καλή κι αν είναι αυτή. Πολλοί πανεπιστημιακοί έχουν ήδη υπογραμμίσει ότι έχουμε ήδη αρκετού κανόνες για την κανονιστική ή νομοθετική διαδικασία. Το πρόβλημα όμως παραμένει σύμφωνα με αυτούς και εξαγούν το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν εφαρμόζονται όλοι οι κανόνε με συνέπεια και συνοχή στην πράξη και γι' αυτό θα πρότεινα να έχουμε ένα ε, ε, σώμα, έναν φορέα κοινό κοινό με εκπροσώπους από τα τρία θεσμικά όργανα και άλλους έτσι ώστε το σώμα αυτό, φορέ αυτό αυτός να είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των κανόνων, με την εποπτεία του πώς εφαρμόζεται αυτοί οι κανόνες. Έχουμε κάποιους κοινούς μηχανισμούς όπως είναι οι τριμερείς διάλογοι, οι τρίλογοι να το πω έτσι και μετά έχουμε και άλλους που ασχολούνται και εποπτεύουν τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ή τη σύνταξη και τη διατύπωση αυτής και του καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή ρυθμίσεις, όμως πρέπει να εξορθολογήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και να έχουν ένα κοινό φορμάτ, μια κοινή ε, μορφή, διαμόρφωση. Είναι καλύτερο αυτό, να έχουμε ένα μόνιμο όργανο, standing body, καλύτερο αυτό από το να έχουμε panel ad hoc επιτόπου. Αυτό, το, το δεύτερο είναι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ε, Συμφωνία για ε, Καλύτερη Νομοθεσία. Better Regulation Agreement. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα πολύ πιο σπουδαίο William Robinson, τον William Heath Robinson και ε, το, η γελιογραφία που βλέπετε στην οθόνη, την οποία έχει φτιάξει αυτός, ε, είναι κάτι που με εμπνέει ιδιαίτερος. Έχουμε πάρα πολλούς εργαζομένους που ε, επιτελεί ο καθένας διαφορετικό έργο και προσπαθούν όλοι μαζί να γεφυρώσουν το, το κενό μεταξύ των δύο πυλώνων και προσπαθούν να φέρουν ένα καινούριο υλικό και νομίζω ότι αυτό το καινούριο υλικό ε, ε, συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο αποτελεσματικό συντονισμό των ε, εργασιών των εμπλεκόμενων, των εργαζόμενων σε αυτή τη διαδικασία είναι αδύρυτη ανάγκη. Δεν θα είναι εύκολο τα τρία θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν πάνω σε ένα κοινό ε, σετ κανόνων για όλες τις τεχνικές πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το αντίθετο μάλιστα, ωστόσο η προσπάθεια πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πάντοτε θα είναι περίπλοκη η διαδικασία, πάντοτε θα είναι δύσκολη η πολιτική διαδικασία, τουλάχιστον όμως. Οι τεχνικοί κανόνες θα είναι πάντοτε σαφείς και θα τους κατανοούν όλοι οι εμπλεκόμενοι αντί να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ε, να τη θεωρήσουμε ως μια χρυσή ευκαιρία να εθετήσουμε μια περιεκτική ολοκληρωμένη συμφωνία για περισσότερες ε, διαστάσεις και πτυχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Ρόμπινσον. Πριν ε, τελειώσουμε την ακρόαση, μήπως υπάρχουν μέλη που θα ήθελαν να σας απευθύνουν ερωτήσεις. Η κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ερώτηση, επιθυμώ όμως να ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και εν ώψη της τόσο σημαντικής και ενδιαφέρουσας αυτής παρουσιάσεως βρίσκω ότι είναι ακόμα περισσότερο κρίμα που είναι απόντες ο κύριος Βεχόφστατ και ο κύριος Τίμερμανς. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κύριε Εμπειρογνώμων για την ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας και ε, σας υπόσχομαι θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα υπέρ μιας βελτίωσης της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ο κύριος Καρίμ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόμπινσον και να του ζητήσω συγνώμη που εκλήθη να εμπλακεί σε μία ευρύτερη συζήτηση. Ζητώ συγνώμη που θα τον ενοχλήσω σε μία δεύτερη φάση. Ε, γιατί νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο ο κύριος Μπερχόφστατ και ο κύριος Τίντερ θα έπρεπε να ακούσουν αυτά που ακούσαμε κι εμείς. Θα ήθελα να ζητήσω επίσης συγγνώμη στους παριστάμενους για την πρόταση που χρειάστηκε να διατυπώσω. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Καρίμ, θα ήθελα να ζητήσω επίσης συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ακρόαση αυτή σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι κύριε Ρόμπινσον. Και θεωρώ ότι λίγη εδώ η ακρόαση, εάν συμφωνεί και η κυρία Ζήμπνερ. Dear colleagues, I just want to say that... Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε συντόμως την συνεδρίαση της Επιτροπής μας.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

Yes. Uh, Θα συνεχίσουμε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι με το υπαριθμόν 16 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για την ε, μετάβαση αντιπροσωπείας στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων που εδρεύει στην πόλη Αλεκάντε της Ισπανίας. Ο κ. Ζβιεύκα. Θα ήθελα Θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία μου ε, σε ό,τι φορά την αποστολή της Επιτροπής Βάσα στο Αλικάντε στην ε, αρχή για την εναρμόνιση εσωτερικής αγοράς. Πήρα, μέρο, πήγα εγώ με την Τερέζα ε, Κομοντίνη και τη Μέρι Χάνιμπολ. Θα ήθελα να πω ότι στην ουσία πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα αποστολή και για τους τρεις μας κυρίως ε, γιατί το πρόγραμμά μας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον από τη στιγμή που μας δόθηκε η ευκαιρία ε, ανεπίσημα να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις προσκλήσεις ε, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο φορέας καθώς και τα προγράμματά του τα οποία είναι σε φάση επεξεργασίας. Θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ στον πρόεδρο και στη γραμματεία και να τους ζητήσω να ετοιμάσουν σύντομα, να προετοιμάσουν σύντομα μία ανταλλαγή απόψεων με τον Διευθυντή κ. Καμπίνος έτσι ώστε ο Διευθυντής να μπορέσει να υποβάλει στην Επιτροπή μας τα ε, προγράμματα του ε, φορέα. Εμείς μιλήσαμε για αυτά τα προγράμματα και πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο όλοι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν γι' αυτό. Θα επιθυμούσα η γραμματεία να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να οργανωθεί μια ανταλλαγή με τον κύριο Καμπύρο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της αποστολής θίξαμε και οικονομικά θέματα και θα, θα πρέπει να πω ότι είναι ο μοναδικός ε, οργανισμός ο οποίος ε, έχει έσοδα, γιατί εκεί καταγράφονται τα, όλα τα σήματα κατά τεθέντα και τα σχέδια. Μιλήσαμε βεβαίως για οικονομικά προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία των διαφόρων οργανισμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση έτσι ώστε αυτό το πλεόνασμα να δαπανηθεί όχι με έναν τρόπο έτσι ώστε να ανακατεταρεμηθεί μεταξύ των διαφόρων ε, γραφείων αλλά προκειμένου να προετοιμαστεί μια δράση κοινοτικού χαρακτήρα δηλαδή που να είναι προς όφελος όλων των χωρών μελών με ένα και να υπάρξει παράλληλα και ένας ε, συνδυασμός του υπεύθυνης υπηρεσίας εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι τον κύριο Καμπίνος θα τον ενδιαφέρε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Μα δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία. Ε, βεβαίως ε, βοηθάει και το πλαίσιο. Το Αλικάντεμι είναι μια πανέμορφη πόλη και συνέβαλε και αυτό. Η έδρα του φορέα της υπηρεσίας είναι στις μεσογειακές ακτές. Ακόμα και σε μια πυρετόδη μέρα εργασίας μπορεί κανείς να σηκώσει το βλέμμα του και να δει έξω το υπέροχο μεσογειακό τοπίο. Τώρα, ας μην χαριτολογούσουμε άλλο, ε, θα ήθελα να πω ότι μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού και αυτό επέτρεψε στον οργανισμό να εφαρμόσει μια διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματική για την διαχείριση των ετοιμάτων. Αυτή η τράπεζα δεδομένων και η διαδικτυακή πόρη που έχει ο οργανισμός επιτρέπει μια άμεση επαφή όχι μόνο με τις χώρες μέλη αλλά και με τις τρίτες χώρες προκειμένου να επαληθευτούν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταγραφή των σχεδίων ένα καλά ρονταρισμένο σύστημα. Για παράδειγμα, είδαμε μία ε, κυρία να εργάζεται σε δύο οθόνες κάνοντας μία προσωμείωση της ε, εγγραφής δύο ε, σημάτων κατατεθέντων. Και η κυρία αυτή μας εξήγησε πως λαμβάνεται η τελική απόφαση εγγραφής. Καταχώρησης, με συγχωρείτε. Ε, αυτό βεβαίως απαιτεί γνώσεις, γνώσεις που τις έχει ο φορέας και οι εργαζόμενοι στον ε, οργανισμό που εγγράφονται στον τομέα των καταχωρήσεων έχουν ε, ειδικέ αίθουσε όπου υπάρχουν οθόνες όπου προβάλλεται το προσυζήτηση αντικείμενο. Δηλαδή κάθε τμηματάρχη σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ελέγξει την όλη διαδικασία εγγραφής μιας ε, καταχώρησης ενός ε, σήματος κατατεθέντος. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για τα παρακάτω θέματα. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων το βράδυ, το ε, και θα έλεγα ότι ήταν και συγκινησιακά φορτισμένη αυτή η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της, ε, του οργανισμού και των ε, ε, βουλευτών. Μας δόθηκε ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο δοσμένοι στη δουλειά τους ήταν οι υπάλληλοι. Μπορέσαμε να δούμε τα διάφορα σήματα, μπορέσαμε να δούμε και τα σήματα γεωγραφικής προέλευσης ενημερωθήκαμε όχι μόνο για την, ε, τις καθημερινές δραστηριότητες ε, του οργανισμού. Μας δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι ε, αποστολές για τα μέλη της Επιτροπής μας. Γιατί στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων μπορούμε να μιλήσουμε και για το μέλλον της νομοθεσίας που μπορεί να αφορά τις εργασίες του ίδιου του οργανισμού. Εμένα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να ευχαριστήσω για αυτή την αποστολή γιατί πραγματικά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Χάνιμπολ. Πολύ σύντομα, ο κύριος Θιεύσκα ήταν ιδιαίτερα επεξηγηματικός. Θα έλεγα ότι ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι, πραγματικά το χαρήκαμε. Όταν ε, δούλευα στο Λονδίνο είχα θέα προς τον Τάμεση, αλλά η θέα ε, προς τη Μεσόγειο είναι ακόμα καλύτερη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να δει κανείς πώς λειτουργεί αυτός ο φορέας. Έχουν ε, πολύ άριθμο προσωπικό, εμείς επισκεφτήκαμε όλα τα τμήματα και όταν μιλάμε για αυτόν τον φορέα δεν καταλαβαίνουμε πόσα πολλά κάνουν και πόσο καλά τα κάνουν. Η όλη η οργάνωση ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Έκαναν κάτι που πραγματικά το βρήκα εντυπωσιακό. Σε κάθε γραφείο είχαν ένα μόνιτορ που ε, ε, έδειχνε τις, εκκρεμότητε τις εκκρεμότητές τους. αγχωτικό λίγο μου φάνηκε. Τώρα, ε, υπάρχει... Ο κύριος Καμπίνος ε, θα επιθυμούσε να έρθει εδώ για να μιλήσει για την εργασία της Επιτροπής. Και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να βρούμε κάποια, ε, ε, κάποιο χρόνο να αφιερώσουμε. Θα έλεγα να κάνουμε μια προσπάθεια. Υπάρχουν προκύπτουν συνέχεια πράγματα και βεβαίως θα γίνουν ε, αλλαγές. Ε, υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Θα έλεγα λοιπόν να οργανώσουμε κάποια στιγμή τη συνάντηση με τον κύριο Καμπίνο. Ναι, συμφωνώ Πήγα στο Αλικάντε πριν από ένα χρόνο για την 20η επέτειο από την ίδρυση του γραφείου και νομίζω ότι θα πρέπει να το προβάλλουμε προς ε, τον κόσμο ως ένα επιτυχές παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ένα στόχο παραπάνω για να καλέσουμε τον κύριο Καμπίνο σε, αυτή την επιτροπή. Πρόσφατα τελειώσαμε με το πακέτο του σήματο καταδεθέντος και θα ήταν χρήσιμο να τον ακούσουμε να μας παραθέτει τι απόψει του σχετικά με την εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού. Ναι, πολύ καλή ιδέα να τον καλέσουμε στη συνάντηση της Επιτροπής μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να περάσουμε στο 17. Αντιπροσωπεία που επισκέπτηκε τον Όσα στο Παρίσι. Η κυρία Ρέγνερ και ο κύριος Ντιράν είναι εδώ. Παρακαλώ, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επίσκεψη στον ΟΣΑ Βεβαίως ήταν πολύ διδακτική. Και φτάσαμε εκεί μάλιστα και σε ένα ενδιαφέρον χρονικό σημείο. Τα θέματα ήταν ευρύτατα, δηλαδή εταιρικό δίκαιο, corporate governance και ιδιαίτερα το θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Το απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για την FPR, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων Το πιο ενδιαφέρον ήταν ε, η συνάντησή μας με τον Άγχελ Γκουρία. Πριν μάλιστα δημοσιευτεί στις εφημερίδες για το G20 και την ε, υιοθέτηση της ε, ρύθμισης για την έκδοση εκθέσεων ανακράτος, αναχώρα και βεβαίως όλα αυτά και εν ώψη του ιστορικού των δικών μας εργασιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρω εδώ την ε, οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και για την corporate governance. Αυτές τις συζητήσεις που δεν κάναμε βέβαια μόνο με τον Γκουρία αλλά και με άλλους επιστήμονες και άλλους υπευθύνους του ΩΣΑ έχω να σας περιγράψω μια εικόνα που μου έμεινε πώς έχουν διαμορφωθεί οι δομές των ιδιοκτητών των μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν χώρες όπου οι κύριοι μέτοχοι, οι οποίοι διαθέτουν ακόμη μεγάλα πακέτα μετοχών, εξακολουθούν να υπάρχουν. Όμως όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις τώρα οι επιχειρήσεις ανήκουν σε όλο και οι υπερτοχές των, των εταιριών δηλαδή, ανήκουν σε ένα όλο και ευρύτερο φάσμα, γιατί οι ήπιες έρχονται συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν σε μετοχές, μετοχών, ε, σε μετοχές σε επιχειρήσεων κ.ο.κ. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετική η εικόνα και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ε, επεκτείνεται και η ευθύνη και για την εφαρμογή των διαφόρων νομοθετικών ε, διατάξεων, δηλαδή για την εκπλήρωση των ε, υποχρώσεων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα ερευνά ο ΩΣΑ και με ένα στόχο να καταστήσει τα πράγματα αυτά περισσότερο δεσμευτικά. Κάναμε και μια συζήτηση με μία από τις βασικότερες ερευνήτριες του ΩΣΑ σε σχέση με το θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, πράγμα το οποίο στηρίζει πολύ όσα και η πρόταση της ερευνήτριας, μάλλον η πρόταση έγινε προς την ερευνήτρια, να προσκληθεί να εμφανιστεί ενώπιόν μας εδώ στην Επιτροπή μας, διότι προβλέπεται και μεγάλη διάσκεψη από την Λουξεμβουργική Προεδρία στο Λουξεμβούργο, στη διάρκεια της Προεδρίας ακόμη, για να θέσει το θέμα και από πλευράς Συμβουλίου. Βρίσκω ότι αυτή η πρόθεση είναι σημαντική, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί ζωντανό το θέμα, αλλά και από πλευράς μας να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση και να ζητήσουμε και περισσότερες πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζει το θέμα όσα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ γιατί ίσως θέλει και ο κ. Ντυρόν να πει λίγα πράγματα. Το Παρίσι δεν είναι μακριά από εδώ, από τις Βρυξέλλες και οι συζητήσεις με τον ΩΣΑ διαμορφώνονται πάντοτε με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο γιατί έχουν και οικονομική και πολιτική σημασία και βέβαια και για τα όσα συμβαίνουν στους G20 τα οποία δεν επιτρέπεται κανείς να υποτιμά. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη στο Παρίσι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εσείς κύριε Ντυρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πια τι να προσθέσω στα πολύ ξεκάθαρα λόγια που είπε η κυρία Ρέγνερ. Ήταν πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ραντεβού. Μέσα στο πρωινό είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αναλύσεις για τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και συγκριτικά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και αυτό έχει ενδιαφέρον διότι βλέπουμε τις τάσεις διαμορφώνται της ΗΠΑ να έρχονται λίγα χρόνια μετά στην Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς βέβαια και το, να συνειδητοποιήσει κανείς και τον αριθμό των διαμεσολαβητών. Δηλαδή ε, έχει ε, εκτοξευτεί πλέον ο αριθμός των μετόχων και κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό και ένα από τα πια μείζωνα θέματα και για τα επόμενα χρόνια. Διότι υπάρχουν και διαμεσολαβητές, οι οποίοι διαμεσολαβητές αμείβονται και αμείβονται αρκετά ικανοποιητικά δικηγόροι που ε, είναι γνωστό ότι αμείβονται καλά, αλλά και οι οικονομικοί διαμεσολαβητές έχουν και επίσης ένα σημαντικό περιθώριο. Και αυτό διαμορφώνει και τις ψήφους και την διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΗΠΑ, αλλά και για τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις που και για παράδειγμα στο 80% ε, στι ΗΠΑ εξαρτώνται από αυτού του είδου τη χρηματοδότηση. Αυτά ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα, καθώ και να τεθεί και το ερώτημα και της ε, ανάμειξης, δηλαδή του, τρόπου που γίνεται η ανάμειξη μέσα στο, στη διακυβέρνηση. Και ο διευθυντής τους είναι πάρα πολύ, σε, φόρμα και η ε, η συνάντηση μαζί του κράτησε διπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλεπόταν και έχει ανάγκη από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το είπε άλλωστε και για το ραντεβού με τους G20. Για τον ΩΣΑ λοιπόν το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, πραγματικό ρόλο και για θέματα βεβαίως δικαιωμάτων των ε, μετόχων και για, την, ε, για τον φόρο επί των συναλλαγών και ούτω καθεξής. Έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να παίξουμε λοιπόν. Ενδιαφέρον λοιπόν ε, ραντεβού, βεβαίω ήταν παρόν και ο κύριο Καβαντά, ήμασταν τρει λοιπόν που πήγαμε και επισκεφθήκαμε τον ΟΣΑ και τον κύριο Γκουρία. Τέσσερι μου φαίνεται, έτσι δεν είναι, λέει ο πρόεδρο. Η Κωνσταντ Λεβί. Ναι, ναι, ε, ε, που με ξέχασα. γιατί όταν ήρθε η Κωνσταντ, εγώ ήμουν υποχρεωμένο να αποχωρήσω για να έρθω να ψηφίσω ο πρόεδρος Φόμποτα. Δεν βλέπω κανείς να ζητεί το λόγο, άρα και αυτό το θέμα ολοκληρώνεται. Η συζήτηση δηλαδή μας μένει ένα θέμα στη μεσαία διάταξη της σήμερα, ο έλεγχος των ε, εκτελεστικών πράξεων με εισηγητή τον κ. χρυσόγων ο οποίος όμως δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή, αλλά από την έκθεση είναι σαφές ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με τις πράξεις αυτές, δηλαδή για την πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για το νομοθέτημα δηλαδή 1126 2000 και το άλλο πάλι το 2002 αυτή τη φορά και το άλλο είναι ε, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί των υπαριθμών 1126 κάθετος 2000 και για την προσαρμογή ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων για να συμφωνούν με τον 1606 του 2000 που αφορά διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αν μπορείτε να τα σημειώσετε αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συζητήθηκε το θέμα. Αν έχετε όμως ερωτήσεις, θα χρειαστεί να το αναβάλουμε για άλλη συνεδρίαση. Δεν έχετε ερωτήσεις? Άρα, εξαντλήσαμε τη σημερινή μας ημερησία διάταξη. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Τελευταία ανακοίνωση, η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται 5η 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλε. Και σας ευχαριστώ πολύ.